Το επόμενο σημείο είναι η έκθεση της κυρίας Ήλτα Φιγκρέντο ε, σχετικά με την ε, κύρωση της σύμβασης του Διεθνού Οργανισμού Εργασίας το 2007 σχετικά με την εργασία στον τομέα της αλίας. Στρέφομαι στην εισηγήτριά μας. Η κυρία Φιγκρέντο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, με αυτή την έκθεση θέλουμε να εγκρίνουμε την πρόταση απόφαση του Συμβουλίου για την Σύμβαση 188 του, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας για την εργασία στον τομέα της αλίας που ορίζει διεθνεί ελάχιστου. Κανόνε και προδιαγραφές που θα πρέπει να γίνονται σεβαστοί, καθώς και συνθήκες περισσότερο ισότιμες σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και το ελάχιστο επίπεδο κύρωση, γιατί, όπως σημαίνει σε πολλέ άλλες συμβάσει και η σύμβαση αυτή που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2007 στην τότε συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασία, όρισε ακριβώ κανόνε και ελάχιστε προδιαγραφέ για τον τομέα τη αλλία προωθώντα αξιοπρεπεί συνθήκε διαβίωσης και εργασία για του εργαζόμενου στον τομέα τη αλίας και τοποθέτηση σε θέματα σημαντικά όπω η ασφάλεια και η προστασία κατά την εργασία, η ώρα ξεκούραση ή στέγαση των αλλιέων, η περίπτωση επαναπατρισμού, μετατόπιση των αλλιών και το κοινωνικό του σύστημα ασφάλισης. Ελπίζουμε στην έγκριση της σύμβασης αυτής ε, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας γιατί θεωρούμε ότι αποτελεί ένα βήμα πρόοδου η σύμβαση για να δοθεί και να κατοχυρωθεί το δικαίωμα εργασίας σε ένα τόσο στρατηγικό εργασιακό τομέα που απασχολεί 30 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι λοιπόν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εργασίας και τα τριμερή όργανα της του οργανισμού αυτού άρχισαν να επεξεργάζονται τις λεπτομέρειες της σύμβασης αυτής για τον τομέα της αλίας προκειμένου να δώσουν στους εργαζόμενους στον τομέα της αλίας ένα ικανό επίπεδο προστασίας σε διεθνές επίπεδο δεδομένων των ιδιαίτερων συνθήκων εργασίας και διαβίωσης των εργαζομένων αυτών που χρειάζεται ειδική ασφάλεια. Μιλάμε για έναν τομέα που προκαλεί και πολλά θανατηφόρα ατυχήματα τα οποία μπορεί να οδηγούν σε περιπτώσεις που να οφείλονται σε περιπτώσεις σοβαρής έλλειψης προστασίας και έλλειψης ασφάλειας. Επίσης η ελάχιστη ηλικία, η ιατρική κατάσταση των εργαζομένων. Η... Το πώς θα, συνθεί, θα συντίθεται το πλήρωμα ενός σκάφους. Όλα αυτά είναι στοιχεία που διέπονται από τη συγκεκριμένη σύμβαση. Έτσι λοιπόν η ενοποιημένη σύμβαση του, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας από τον Φεβρουάριο του 2006 θα έρθει να συνδυαστεί με αυτήν την σύμβαση. Θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλα τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν στην ταχεία κύρωση της σύμβασης κατά προτίμηση πριν το 2012 καθότι η σύμβαση αυτή θα έχει σοβαρά αποτελέσματα, ιδίω εάν ε, κυρωθεί από 10 τουλάχιστον από τα 180 κάτι μέλη της, ε, του Παγκόσμιου Οργανισμού εργασία, εκ των οποίων 8 θα πρέπει να είναι παράκτια. Θα πρέπει κατεπηγόντω να ε, υλοποιηθούν οι διατάξεις της σύμβασης, όπου δεν συμβαίνει ήδη αυτό. Ελπίζω θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όσους βοήθησαν στην επεξεργασία του έκθεση αυτή, περιλαμβανομένου του κυρίου Βίλι Μάγερ, που είναι και μέλο τη Επιτροπή Αλίας Και ελπίζω οι κυβερνήσει και οι υπεύθυνοι των κρατών μελών, ε, οι αρχικοί κρατών και κυβερνήσεων, να προχωρήσουν στην γρήγορη κύρωση τη σύμβαση αυτή. Ευχαριστώ και τώρα Επίτροπο Σπίτλα αξιότιμοι βουλευτές, η αλληλεία εξορισμού είναι ε, παγκοσμιοποιημένος κλάδος και άρα πλήττεται και από την παγκοσμιοποίηση σε μεγάλο βαθμό. Απασχολούνται 30 εκατομμύρια άνθρωποι σε αυτό τον κλάδο οι οποίοι εκτίθενται στους κινδύνους της παγκοσμιοποίησης, ε, αλλά και σε πολλούς ε, κινδύνους, σε πολλά δεινά. Όταν ε, μιλάμε για θανατηφόρα ατυχήματα στον κλάδο της αλίας, με ένα ποσοστό θανατηφόρων ατυχημάτων, εργασιακών ατυχημάτων, πολύ υψηλό βάσει των στοιχείων του, του Διεθνού Οργανισμού Εργασίας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι είναι από τα πιο επικίνδυνα επαγγέλματα στον κόσμο. Όλοι υποστηρίζουν το ε, παγκόσμιο πρόγραμμα σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία στον κλάδο αυτό. Εμείς ενισχύσαμε τη δέσμευσή μας μέσα από μια κοινωνική ατζέντα και μια ανακοίνωση για την αξιοπρεπή εργασία το 2006. Υποστηρίζουμε ε, τα διεθνή πρότυπα σε αυτό το τομέα και ε, βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης ε, καθώς και της νομικής προστασίας ε, που παρέχεται στους εργαζομένους. Όλα αυτά ε, θα γίνουν εφικτά μόνο αν τηρηθούν τα διεθνή πρότυπα. Ως μέλη στο Διεθνή Οργανισμό Εργασίας ε, συμβάλαμε και εμείς ε, στην ε, επικαιροποίηση αυτής της σύμβασης όπου θεσπίζονται ελάχιστα πρότυπα για την αξιοπρεπή εργασία και θεσπίζονται και κάποιοι μηχανισμοί για τις επιθεωρήσεις που γίνονται στους λιμένες πέρα από αυτή τη σύμβαση που δεν είναι νομικά δεσμευτική και να πω εδώ παρενθετικά το τον Ιούνιο του 2007 εγκρίθηκε αυτή η σύμβαση από την ε, Διευθυντική Επιτροπή του Διεθνού Οργανισμού Εργασίας. Πρόκειται για σύμβαση 188 χάρη στην οποία θα υπάρχουν οι ίσες συνθήκες εργασίας ε, για όλους, ε, ρυθμίζονται θέματα όπως ε, το ελάχιστο ηλικιακό όριο, ο ιατρικός έλεγχος, ο χρόνος ανάπαυσης του πληρώματος, συμβάσεις εργασίας, ο επαναπατρισμός, η πρόσληψη των εργαζομένων, ο μισθός τους, η σύντηση, η ενδιέτηση, η κοινωνική ασφάλιση. Ε, η σύμβαση εν μέρη σχετίζεται και με την εναρμόνιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Ε, αυτό είναι αμυγός κοινοτική αρμοδιότητα. Γι' αυτό και το Συμβούλιο θα πρέπει να επιτρέψει στα κράτη-μέλη να επικυρώσουν αυτά τα συγκεκριμένα τμήματα της σύμβασης ε, του ΔΟΕ υπάρχουν και κάποια άλλα τμήματα που σχετίζονται με άλλα θέματα. Υπάρχει ένα νέο πρότυπο Υπάρχουν νέα πρότυπα, μάλλον θεσπίστηκαν από τον ΔΟΕ, που θα αρχίσουν να ισχύουν μελητεί, Οπότε προτείνει η Επιτροπή μέσα αυτή τη σύμβαση να συμπεριλάβουμε μία έκκληση προ τα κράτη-μέλη, ούτω ώστε το ταχύτερο δυνατόν να επικυρώσουν την σύμβαση ή δυνατόν μέχρι το Δεκέμβριο του 2012. θα γίνει έλεγχος από το Συμβούλιο μέχρι τον Ιούνιο του 2012 σε σχέση με την επικύρωση αυτής της σύμβασης. Σας ευχαριστούμε. Και τώρα χωριτές εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Πρώτος ο κύριος Μπραγκέτο εκ μέρους του ΕΛΚ για τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ επίτροπε. Όπως γνωρίζουμε, αλλά όπως και υπόθηκε απόψε, ο τομέας της αλίας θεωρείται από τον ΔΟΕ ως ένας από τους τομέας, τους τομείς εργασίας τους πλέον επικίνδυνες. 24.000 θανατηφόρα ατυχήματα ετησίως. Σας δείχνει αυτό τι διαστάσεις μπορεί να λάβει αυτό το πρόβλημα. Είναι ένας τομέας όμως ο οποίος πρέπει να υπόκειται σε, και υπόκειται σε διεξοδικούς διεθνείς κανόνες προκειμένου όμως να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και προστασία στους εργαζομένους του τομέα σε όλο τον κόσμο. Πολλέ φορέ μάλιστα είναι αντικείμενο εκμετάλλευση εργαζόμενου αυτή. Η Σύμβαση 188 για τον εργασία στον τομέα τη Αλία είναι θεμελιώδου σημασία. Θέλει να ορίσει ισότιμε συνθήκε εργασία και δικαιότερου όρου ανταγωνισμού για τον εν λόγω τομέα ε, αφορά την αξιοπρεπή εργασία και διαβίωση των ναυτικών, των εργαζομένων στον τομέα της αλίας, καθώς και την σύνθεση του πληρώματος, την ιατρική περίθαλψη, την αμοιβή, την κοινωνική ασφάλεια. Όλα αυτά τα στοιχεία που προαναφέρθησαν σε σχέση με τους εργαζόμενους στο τομείο της αλίας. Υπάρχει λοιπόν συμφωνία εδώ για τη σημασία των κανόνων αυτών και το μόνο που θέλω είναι να τονίσω την ανάγκη και το κατεπήγον να προχωρήσουμε σε κύρωση, κύρωση της σύμβασης από τα κράτη-μέλη, ώστε να ελοπιθούν και εν λόγω κανόνες όσο το δυνατόν συντομότερα. Ευχαριστώ. Και τώρα εκ μέρους των σοσιαλιστών ο κύριος Ντερόσα για τρία λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο που μπορώ να μιλήσω για αυτό το ζήτημα εδώ απόψε. Διότι νομίζω ότι η δουλειά ενός ψαρά ή μιας γυναίκας που δουλεύει και εκείνη σε ψαράδικο είναι από τις πιο επικίνδυνες στον κόσμο. στην Ιρλανδία πέρσι μόνο πάνω από ένα σκάφι χάθηκαν στη θάλασσα. Είναι αρκετά τα σκάφη που χάθηκαν στη θάλασσα και πολλοί είναι αυτοί που τραυματίστηκαν στον τομέα της αλίας, άνδρες και γυναίκες. Λες και είχαν πάει στον πόλεμο. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να καλύψουμε στην Ιρλανδία τα δικαιώματα των ανθρώπων που εργάζονται σε αλλιευτικά σκάφη. Μιλάμε για ένα τομέα ιδιαίτερα περίπλοκο. Διότι σημαντικό είναι με τι είδου σύμβαση εργάζεται ο εργαζόμενος κατά πόσο είναι τακτικοί εργαζόμενοι και κατά πόσον ε, έχουν, καταβάλουν τις εισφορές τους σε ένα ταμείο ή στον ε, καπετάνιο του πληρώματος ή αυτόν ο οποίος είναι υπεύθυνο για τα αλλιεύματα. Εφόσον δεν είναι και τακτικοί εργαζόμενοι. Το να συμφιλιώσουμε λοιπόν όλες αυτές τις διαφορετικές κατηγορίες και περιπτώσεις είναι εξαιρετικά πολύ σύνθετο. ως υπουργό. Είχα εντοπίσει μάλιστα ένα ευρωπαϊκό νομοθέτημα που είχε δημιουργήσει προβλήματα. Ευτυχώς βραχυπρόθεσμα. διότι ακριβώ δεν μπορούσε να ισχύει απολύτω ω εργασιακό δίκαιο για την εν λόγω εργασιακό τομέα. Χρειάζονται λοιπόν ελάχιστα πρότυπα και προδιαγραφές. Ε, είναι αναγκαίο αυτό η ιατρική περίθαλψη, η διαβίωση των ναυτικών, η σύντησή τους, η ελάχιστη αμοιβή του, όλα αυτά τα ζητήματα είναι αναγκαία για του εργαζόμενου στον τομέα τη Αλίας Υπάρχει λοιπόν υποχρέωση και από τους πλειοκτήτε και από τους ε, καπετάνιους του πληρώματο να βεβαιωθούν ότι καταβάλλονται τα δέοντα στους εργαζομένους. Αλλά τα ελάχιστα αυτά πρότυπα απαιτούνται διότι υπάρχουν και τάσεις να μειώνονται όσα οφείλονται στους εργαζομένους. Τάση που υπάρχει και σε άλλους τομείς βεβαίως. Πρέπει λοιπόν να αναχαιτήσουμε αυτή την τάση όσο το δυνατόν συντομότερα. Γι' αυτό παροτρύνω να κάνουμε τα πράγματα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μπορούμε. Το 2012 είναι μακριά ή δυνατόν να συντομεύσουμε τις διαδικασίες κύρωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ιντεμ, κυρία Σίνοτ, δύο λεπτά. Είναι πολύ σημαντικό οι αλληλείς να έχουν συνθήκες εργασίας λογικές, ασφαλείς, γιατί είναι υψηλού κινδύνου ε, επάγγελμα η δυνατον να συντομευσουμε τις διαδικασιες σας ευχαριστω ευχαριστω ιντεμ κυρια σινοτ δυο λεπτα ειναι πολυ σημαντικο οι αλληλεις να εχουν συνθηκες εργασιας λογικες ασφαλεις γιατι ειναι υψηλου κινδυνου επαγγελμα η αλληλεια οι άνδρες και οι γυναίκες πρέπει να μπορούν να υποστηρίζουν τον εαυτό τους, την οικογένειά τους και επίσης θα πρέπει το εισόδημα να είναι σταθερής βάσεως ούτως ώστε να παραμείνει η παράκτια κοινότητά τους. Οι παράκτιες κοινότητες ε, δύσκολα επιβιώνουν στη χώρα μου τουλάχιστον. Το θέμα για μένα είναι αν η κύρωση της 188 σύμβασης του Ισδόε θα επεκτείνοντας ε, τη, τους κανόνες ε, στους αλληλείς θα αποτελέσει εμπόδιο η προστασία για, για τους αλληλείς. Θα μπορέσει να ε, εξασφαλίσει ίσως κανόνες του παιχνιδιού για να επιβιώσουν γιατί οι προϋποθέσεις εργασίας και οι συνθήκες εργασίας δεν είναι καλές. Γνωρίζω ότι η αλληλεία ε, πολλές φορές δεν ωφελεί τρίτες χώρες ε, και οι συμβάσεις ε, που έχουν συναυθεί δεν τους καλύπτουν. Στην Ιρλανδία οι αλληλείς που δεν έχουν δουλειά δεν καλύπτονται από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Αν η κύρωση λοιπόν ε, αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά, κοινωνική ασφάλιση, ανεργία, ε, οικονομική βιωσιμότητα, τότε τη χαιρετίζω. Καλό είναι η αλία να είναι βιώσιμη και για τις μικρές κλίμακας αλίες τότε. Ναι, γιατί ούτως ή άλλως η αλία ελια ειναι επικίνδυνη και πολλές φορές ε, το αντικείμενο εκμετάλλευσης ε, δεν είναι τα ψάρια μόνο, αλλά και οι ίδιοι οι αλίες. Εξ ονόματος των μη εγγεγραμμένων, ο κύριος Μαρτίνες, δύο λεπτά. Πρόεδρε, Επίτροπε, η αηφόρος διαχείριση της αελίας συνεπάγεται φυσικά αύξηση των ελεγχών, αλλά επίσης θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες και οι αηλίες. Όταν μιλάμε ε, για την αιλία όλοι γνωρίζουμε ότι είναι το ε, πλέον δύσκολο επάγγελμα, παρότι έχει εξελιχθεί η κατάσταση από το 19ο αιώνα, φεύγαν οι Ιρλανδοί και πηγαίναν στα πέλαγα, ε, αλλά όλοι γνωρίζουν τους κινδύνους κινδύνους ε, και τις δυσκολίε του επαγγέλματο. Ε, λόγω τη ε, παγκοσμιοποίηση και τη παγκοσμιοποίηση των αλλιευτικών πόρων, οπωσδήποτε πρέπει να είναι διεθνή και τα πρότυπα. Και φόσον δεν μιλάμε για διεθνή ρύθμιση του επαγγέλματος. Λόγω της παγκοσμιοποίησης και της παγκοσμιοποίησης των αλλιευτικών πόρων οπωσδήποτε πρέπει να είναι διεθνή και τα πρότυπα. Και εφόσον δεν μιλάμε για διεθνή ρύθμιση του επαγγέλματος, ο νομοθέτης δεν μπορεί να είναι παρά ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας και ναι, είναι και η πεντηκοστή επέτειο εξάλλου των συμβάσεων του ΔΟΕ για διάφορα ζητήματα, για την ένδυση, συγγνώμη, τη σύντηση, την ενδιέτηση ε, και άλλα τέτοια ζητήματα και γι' αυτό ε, ο ΔΟΕ τώρα αναθεωρεί διάφορες ε, συμβάσεις και φυσικά μέχρι το 2010 θα πρέπει να επικυρωθούν αυτές οι συμβάσεις από τα κράτη-μέλη. Βλέπουμε ότι πρόκειται για κοινού παγκόσμιου πόρους και θα πρέπει να τους διαχειριστούμε από κοινού γιατί υπάρχει πολύ ισχυρό ανταγωνισμός και υπάρχουν πολλές καταχρήσει στον κλάδο της αλληλεία. υπάρχει εκμετάλλευση, ε, θα έλεγα και σκλαβιά ε, για να μειωθεί το κόστος. Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρξει νομοθετική προστασία για το χρόνο εργασίας, ε, για τις συνθήκες εργασίας, για τους μισθού, για την υγειονομική περίθαλψη, για τη σύντηση, για την ενδιέτηση και την ασφαλιστική κάλυψη. Εδώ έχουμε ένα, μια μήνυμη σε νομοθετική ρύθμιση για τους αλείς για να αντιμετωπίσουν τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Ε, οι Ευρωπαίοι αλείς ε, ήδη έχουν προστασία, αλλά για τους αλείς από το Περού, παραδείγματος χάρη από την Αφρική, αυτό συνιστά μεγάλη πρόοδο. Ευχαριστώ. Ε, μεμονωμένοι ομιλητέ. Ε, πρώτη κυρία Παναγιωτοπούλου Κασιό του. Τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, θεωρώ πολύ σημαντική την ε, απόψινή συζήτηση γιατί ε, με την συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με το ψήφισμα που θα υποστηρίξουμε όλοι ομοφόνος φαντάζομαι αύριο, θα δώσουμε ακόμα μία όθηση στην πραγματοποίηση της ατζέντα αξιοπρεπούς εργασίας, την οποία όλοι μαζί υποστηρίξαμε πέρσι, γιατί η Σύμβαση 188 δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα κομμάτι της εφαρμογής αυτής της ατζέντα στον ε, τομέα της αλληλείας, ο οποίος δεν καλύφθηκε από την ενοποιημένη σύμβαση για την ναυτική εργασία ε, και ε, όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές είναι πολύ σημαντικό και στον τομέα αυτό να έχουμε μια ελάχιστη κάλυψη σε παγκόσμια κλίμακα. Ε, οι χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης φαντάζομαι ότι θα επικυρώσουν όλες όπως προβλέπεται μέχρι το 2012 τη σύμβαση αυτή άλλωστε 8 κράτη μέλη έχουν όλες επικυρώσει άρα η σύμβαση θα αρχίσει να ισχύει και έτσι θα ε, μπορούμε να ε, είμαστε υπερήφανοι όσοι κατοικούμε στα παράλια ότι ε, οι ναυτικοί μας, οι αλληλείς μας θα έχουν κάλυψη αλλά δεν θα έχουν και ανταγωνισμό από τις τρίτες χώρες οι οποίες θα μπορούν να έχουν ε, υποστήριξη κοινωνική για τους αλληλείς τους. Ε, να θυμίσω ότι το Κοινοβούλιο έχει κιόλας ε, ψηφίσει υπέρ της προστασίας και των γυναικών που ασχολούνται ή που έχουν σχέση με την αλληλεία και είναι πολύ σημαντική η ενασχόληση των γυναικών με την αλληλεία είτε έμεσα είτε άμεσα γιατί αν δεν ήταν πίσω από τους αλληλείς ε, οι γυναίκες των ε, παράκτιων περιοχών ε, θα ήταν πολύ φτωχότερες και πολύ λιγότερο καλυμμένες γιατί την κάλυψη στις ανάγκες την κάνουν οι άνθρωποι και όχι μόνο τα νομοθετικά κείμενα. Συμβάλλουμε λοιπόν σε ένα πολιτισμό των παράκτιων περιοχών πολιτισμό κοινωνικό κοινωνικό ε, που ε, θα αξιοποιήσει τα πολιτιστικά στοιχεία της Ευρώπης δεμένα με τη θάλασσα και τις παράκτιες περιοχές από το νότο μέχρι το βορρά. Ε, κάθε περιοχή έχει τις ιδιαιτερότητές της, όμως ε, η σύμβαση που ε, αποφασίζουμε να κυρωθεί από τα κράτη-μέλη δίνει κάλυψη για κάθε περίπτωση και κάθε ανάγκη των αλλιέων. Ιδιαίτερα ε, πρέπει να ε, υποστηρίξουμε ότι θα πρέπει να ε, ληφθεί μέρημνα και για την εκπαίδευση και την εξασφάλιση των γυρατιών τους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Πάμε στο κομμάτι Catch the Eye. Η κυρία Ροϊτόβα έχει ζητήσει πρώτο λόγο. Επίτροπε, όπως και οι συνάδελφοί μου, Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να εγκριθούν πρότυπα που θα εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους εργαζομένους στον τομέα της Ιαλίας. Στον 21ο αιώνα είναι απαράδεκτο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υφίστανται ακόμη συνθήκες εργασίας που προσωμιάζουν τη σκλαβιά. Ε, χαίρομαι ιδιαίτερα που εγκρίθηκε αυτή η προσέγγιση από τα ε, τα τριμερή όργανα του ΔΟΕ, δηλαδή οι εργοδότες, ε, ε, οι εργαζόμενοι και οι κυβερνήσεις, ε, οι εθνικές αρχές. Έτσι ορίζονται το ελάχιστο ηλικιακό όριο, οι ιατρικές επισκέψεις, ο χρόνος ανάπαυσης, η κοινωνική ασφάλιση και άλλα ζητήματα, χάρη στα οποία θα έχουμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας πλέον για τους αλλοίς. Ε, εμείς δεν έχουμε, ε, δεν, βρέ, δεν βρέχει τη χώρα μου από θάλασσα, αλλά τέλος πάντων παρόλα αυτά χαίρομαι πάρα πολύ που εξασφαλίζεται έτσι η προστασία των εργαζομένων και ζητώ την ταχύτατη ε, κύρωση των συμβάσεων. Βέβαια μου αρέσει πολύ το ψάρι αν αυτό βοηθάει. ευχαριστούμε ο κύριος Καζάκο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ενώσω τη φωνή μου με τη φωνή της εισηγήτριας του Επιτρόπου όλων των συναδέλφων που εξέφρασαν την ευχαρίστησή τους, την ικανοποίησή τους για αυτήν την σύμβαση του ΔΟΕ και βεβαίως την ανάγκη όλα τα κράτη-μέλη να κυρώσουν την εν λόγω σύμβαση. Το θέμα εδώ για την αγορά αυτή του τομέα αλίας που δεν είναι ακόμα εναρμονισμένος, δεν είναι ρυθμισμένος, είναι μια άγρια ζούγκλα. Αυτό έχει συνέπειες και για τους ε, καταναλωτές και για τους αλίες, αλλά και για τον ίδιο τον εργαζόμενο στον τομέα αλίας. Διότι ο Αλιεύ θα πρέπει να είναι αυτό που θα βρίσκεται στο κέντρο τη κοινή αλλιευτική πολιτική. Αυτό είναι το σημείο αφετηρία. Δεν θα πρέπει να μείνουμε στην κύρωση, την απλή κύρωση τη διεθνού αυτή σύμβαση, αλλά θα πρέπει να βάλουμε στο κέντρο τη κοινή μα αλλιευτική πολιτική τη ζωή και τον ίδιο τον Αλιέα, τον ψαρά. Ευχαριστώ και τώρα στρέφομαι στον Επίτροπο, κύριε Σπίτλα. Πρόεδρε, ε, Αγαξιότιμοι βουλευτές, ε, θα ήθελα να σας πω ότι Χαίρομαι ιδιαίτερα που συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση και άκουσα όλα τα, όλη την επιχειρηματολογία των βουλευτών, γιατί έτσι τονίζουμε ακόμη περισσότερο τη σημασία αυτής της σύμβασης, που είναι και το αντικείμενο της ε, ε συζήτησής μας. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η σύμβαση για την καθημερινή ζωή ε, των εργαζομένων στον τομέα της αλίας. Σας είπα ότι αριθμεί 30 εκατομμύρια εργαζόμενους ε, ο κλάδος αυτός. Είναι σαφέστατη η επίσημη διαδικασία επικύρωσης ε, της σύμβασης, οπότε θα πρέπει πολιτικά να κατευθυνθούμε προς την ταχύτατη κύρωση ε, της σύμβασης. Αυτή η ημερομηνία που προανέφερα είναι η καταληκτική ημερομηνία. Ε, καλό θα ήταν να επικυρωθούν και ταχύτερα οι συμβάσεις. Ευχαριστώ την εισηγήτρια, την κυρία Φιγκυρέντο και ευχαριστώ όλους τους βουλευτές για την υποστήριξή τους. Ευχαριστούμε, Επίτροπε. Και τώρα η κυρία Φιγκέιρα εδώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τον Επίτροπο και όλους τους συναδέλφους βεβαίως που παρενέβησαν για να στηρίξουν και να συμφωνήσουν με την κύρωση της σύμβασης αυτής. Βεβαίως, αύριο η έκθεση θα εγκριθεί από το Ευρωκοινοβούλιο, οπότε έτσι θα συνεισφέρουμε κι εμείς όπως δει, ώστε η σύμβαση 188, συνοδευόμενη από την 199, ε, θα εγκριθεί, να εγκριθεί μάλλον σύντομα από τα κράτη-μέλη. Όπως εδώ υπόθηκε, στόχος μας είναι να τεθεί σε ισχύ ως το δυνατόν συντομότερα ή δυνατόν πριν από το 2012 διότι θέλουμε να πετύχουμε τον απόλυτο στόχο τη ε, κύρωση από όλα τα κράτη-μέλη. Θα υπάρχουν έτσι ελάχιστοι κανόνε και σε διεθνή επίπεδο που θα εγγυώνται περισσότερη ασφάλεια και καλύτερε συνθήκε εργασία για του αλληλεί, καθώ και λιγότερα θανατηφόρα ατυχήματα. Σε ένα τομέα που είναι πολύ επικίνδυνο, αλλά και στρατηγικής σημασία. Επίση, θα συνεισφέρουμε κατά τον τρόπο αυτό για να βελτιώσουμε την αξιοπρεπή εργασία των ε, αλλιέων οι οποίοι κάνουν μια τόσο δύσκολη και σκληρή δουλειά και θα πρέπει να βρισκόνται στο κέντρο των μεριμνών και ανησυχιών μα. Σας ευχαριστούμε. Η συζήτηση έχει κλείσει. Η συνέχεια αύριο στις 14 Ιανουαρίου 2009 από τις 9 το πρωί έως τη 1 και μετά από τις 3 ως τις 8 και από τις 9 έως τα μεσάνυχτα. Η ημερή διάταξη είναι δημοσιευμένη και στο ίντρανετ. Κυρίσω τη λήξη της συνεδρίασης.